Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσει η συνεδρίαση της ε, επιτροπή Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ανάπτυξης και, και Προϋπολογισμού. Εξ ονόματος των τριών Προέδρων θα ήθελα να σας καλωσορίσω Ήρθαμε στην έδρα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλώς ήρθαν ε, ε, λοιπόν όλα τα μέλη των τριών επιτροπών. Για τρίτη φορά συνεδριάζουμε σε κοινή επιτροπή για να εξετάσουμε την πρόταση δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ε, εξωτερικού σχεδίου επενδύσεων. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΑΦΕΤ που μας φιλοξενεί σήμερα. Η διαδικασία αυτή της κοινή επιτροπής ε, δημιουργεί αρκετές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, οι συγητές, ο κ. Κούκαν που εκπροσωπείται από την κυρία Μανέσκου, ο κύριος Φρουντζούλιτσα και η κυρία Κάρδια Ζαμπάρη, είναι τρεις συγητές που κατόρθωσαν να συνεργαστούν και να μας παρουσιάσουν το σχέδιο έκθεσης, το οποίο διαμόρφωσαν μέσα σε πνεύμα συνεργασίας. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 24 Τρίτου Παρασκευή στι 12 το μεσημέρι και θα τεθεί σε ψηφοφορία το σχέδιο στι 24 Απριλίου. Η Επιτροπή προπολογισμών βρίσκεται σε ε, ιδιάζουσα κατάσταση διότι μαζί με άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ εξετάζει εκ παραλίλου αρκετές ε, προτάσει που έχουν άμεση σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του ΕΦΣΥ το οποίο ενέπνευσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το, το Ταμείο ELM, καθώς ε, και η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, που δημιουργεί ένα κοινό ε, ταμείο καταβολής είναι όλα θέματα τα οποία εξετάζουμε. Θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι ε, συνεπή όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουμε για τις συζητήσεις των διαφόρων ε, μέσων και σχεδίων. Και τούτου λεχθέντος θα δώσω το λόγο στους συμπροέδρους μου, ίσως την κυρία Λίντα Μακάβαν, καταρχήν. Ευχαριστώ. Κοίτα, δεν θα πω τίποτα. Μπορούμε να ακούσουμε τους συνεισηγητές και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Γιατί συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν. Ο κ. Άντερς Φίτισεν, εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλωσορίζω όλους σας στην τρίτη αυτή κοινή συνεδρίαση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη μετά από ανταλλαγή απόψεων του Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και την ε, συζήτηση με του διάφορου εμπειρογνώμονε και του εμπλεκόμενου φορεί. Θα συζητήσουμε το κοινό προτείνουμε τρει εισηγητέ. Λοιπόν, αυτό το ταμείο τη προτάσεω είναι βασικό στοιχείο για το πενετικό σχέδιο που θα καλύψει τα ριζικά αίτια τη μετανάστευση και θα προωθήσει τι επενδύσει στην Αφρική και στη γειτονιά. Θέλουμε να αυξήσουμε τι ανταποκρίσει στι μεταναστευτικέ πιέσει, μακροπρόθεσμα και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Αυτό το Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη θα δώσει καινοτόμε λύσεις επιτόπου και εστιάζεται επί αναπτύξεω του ιδιωτικού τομέα. Ευπρόσδεκτο αυτό. να εξασφαλίσουμε ε, την επίτευξη της αξίας και καλύπτεται το κενό στο φάσμα διαθεσίμων μέσων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Προσβλέπουμε στις απόψεις των ε, συνεισηγητών που προσπαθούν να τροποποιήσουν αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Μακάγωνα τώρα θα προεδρεύσω των παρεμβάσεων. Θα ξεκινάμε από τους συνεισηγητές. Έξοχη δουλειά, έξοχη συνεργασία. Δύο μεγάλες επιτροπές, μια μικρότερη, Είχαν πει στην αρχή θα είναι δύσκολα, αλλά πήγαν πολύ καλά. Η κυρία Μανέσκου ξεκινά, που αντικαθιστά τον κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω τις σημειώσεις του κυρίου Κούκαν. Ζητά συγγνώμη που δεν παρίσταται. Αλλά θα διαβάσω. Ο εισηγητής καλωσορίζει την καλή συνεργασία με τους εισηγητές των άλλων επιτροπών εν του σχεδίου εκθέσεως εκ μέρους της ΑΦΕΤ θέλει να υπογραμμίσει τον κοινό στόχο δημιουργία ενό οικονομικού μέσου που θα τονώσει τι επενδύσει του ιδιωτικού τομέα στην Αφρική. Και στην ευρύτερη γειτονιά θα προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και θα εκριζωθούν τα, κάποια τα βασικά αίτια τη μεταναστεύσεω. Τονίζει επίση ότι βασικό πρόβλημα είναι να τονώσουμε την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, κυρίω στι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε, για να επιτευχθεί ο λόγο στόχο χρειάζονται και τρεις πυλώνες του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου να συντονιστούν και επενδύσεις μπορεί να επιτύχουν μόνο αν στηριχθούν από την τεχνογνωσία μας, την τεχνική αρρωγή και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος της χώρας εταίρους. Λοιπόν, αυτό το ταμείο είναι μια νέα οικονομική συνιστόσα του σχεδίου για τις εξωτερικές επενδύσεις. Η φιλοδοξία μας είναι να ξεπεράσουμε τα εφιστάμενα μέσα, στηρίζοντα καινοτόμε χρηματοδοτήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω μοντέλων. Αυτό πρέπει να τονώσει αυτό το νέο ταμείο να γίνουν επενδύσεις εκεί που άλλα οικονομικά μέσα αποτυγχάνουν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε επακριβώ και σωστά την αρχή τη προσθετικότητα. Ε, η οποία είναι στην καρδιά του μέσου που προτείνεται το μέσο. Αυτό θα πρέπει να εντοπίζει δυνατότητες επενδυτικές σε διάφορους τομείς στις αναπτυξιακές χώρες και να κατευθύνει τις εγγύσεις οικονομικές σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Φιλοδοξία μας είναι να προσελκύσουμε και ιδιωτικούς επενδυτές για αυτές τις προσπάθειες. Για να το πετύχουμε αυτό θα χρειαστούμε αρκετή ευελιξία, ανοιχτή προσέγγιση, αποτελεσματική συνεργασία με διάφορους ε, διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς Επίσης όμως χρειαζόμαστε σαφείς πολιτικές κατευθύνσεις. Γι' αυτό στο σχέδιο εκθέσεως προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη δομή διακυβερνήσεως του Ταμείου αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου του Κοινοβουλίου και θέλουμε να έχουμε καλύτερα κριτήρια επιλεξιμότητα και καλύτερη δυνατότητα ελέγχου. Το νέο αυτό μέσο προτείνεται, μπορεί να είναι επιτυχέ, εάν δεν το υπερφορτώσουμε με διάφορε προτεραιότητε. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δημιουργούμε ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να τονώσει την ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα, έτσι συμβάλλοντας η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη στι αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι φιλόδοξο στόχος, μακροπρόθεσμο εγχείρημα, γι' αυτό θα είναι σημαντικό να έχουμε σαφείς στόχου και προτεραιότητες ευθύ εξ αρχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Φρουτσουλίκα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλο προνόμιο που μπόρεσα να συνεργαστώ με τους συναδέρφους από την ΑΦΕΤ και την Επιτροπή Προπολογισμών και εκφράζω την ικανοποίησή μου για το αποτέλεσμα. Οι κύριες ανησυχίες μου, πώς θα συμπεριληφθούν τα κριτήρια DAC, της Επιτροπής δηλαδή Αναπτυξιακής ε, Αρρωγής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα, ε, φοροδιαφυγή, έχουν συμπεριληφθεί. Έχουμε κάποιες τροπολογίες προκειμένου να αντικατοπτριστεί η άποψή μα καλύτερα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι ο κύριος στόχος του Ταμείου αυτό, του ΕΤΘΑ, είναι η απάλληψη της φτώχειας και μείωση των ανισοτήτων. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί και το μεταναστευτικό. Γι' αυτό πρέπει με τη βοήθεια του Ταμείου αυτού να έχουμε περισσότερες επενδύσεις σε πιο ευάλωτε χώρες την κατανομή θα τη δούμε όσον αφορά την ενέργεια, το κλίμα, για να ανταποκριθούμε στα όσα υποσχεθήκαμε στο Παρίσι. Πρέπει να υπογραμμίσουμε επίσης τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έχουν πρόσβαση έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις χώρες εκείνες όπου τέτοια χρηματοδότηση είναι πρόβλημα. Η μεικτή συνελευσία και Ευρωπαϊκή Ένωση λογοδοτεί στις χώρες μέλη και τους πολίτες. Οπότε η εγγύηση αυτή επενδύσεων μπορεί να βοηθήσει τις χώρες εταίρους. Χαίρομαι που στην έκθεση λέει ότι το Ταμείο αυτό δεν θα βοηθήσει χρηματοδότηση δράσεων που έχουν να κάνουν με την άμυνα, την ασφάλεια, τους εξοπλισμούς ούτε θα στηρίξει ενεργειακά προγράμματα που περιλαμβάνουν τα πυρηνικά. Επειδή υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στις χώρες εταίρους. Ή άλλες επενδύσεις που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις χώρες εταίρους. Κατά του περιβάλλοντος εκεί δηλαδή ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Προσβλέπω στην συνεργασία μας για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Καρδιά τώρα. Από την Επιτροπή Προπολογισμών. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε, είχαμε εξαιρετική συνεργασία οι τρεις συζητητές. Τα πάνε εκείνοι, οπότε λίγα με να προσθέσω εγώ. Όμως κάποια γενικά σχόλια θέλω να κάνω για το πνεύμα μέσα στο οποίο συνεργαστήκαμε. Όπως είδατε, συμφωνούμε σε ένα μεγάλο βαθμό με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θελήσαμε σε κάποια σημεία της πρότασης να μπούμε περισσότερο σε λεπτομέρειες και να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα που θεωρούσαμε ότι δεν αναφέρονταν επαρκώς. Όσον αφορά το στόχο, συμφωνούμε απόλυτα. Θέλουμε όντω να ενισχύσουμε τι επενδύσει στι χώρε που βρίσκονται γύρω από εμά, στο βορρά, στον νότο, στην Αφρική και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό μέρο του ευρωπαϊκού προπολογισμού να το χρησιμοποιήσουμε σαν εγγύηση για να δώσουμε κίνητρο και να προσελκύσουμε νέε επενδύσει. Με μειωμένο συνεπώ κίνδυνο. Υπάρχουν τρει πυλώνε. Ο ένας είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά δίνουμε την ίδια σημασία και στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα που δεν αποτελούν μέρος του κανονισμού πάνω στον οποίο δουλέψαμε, αλλά θελήσαμε να αναφερθούμε και στους δύο άλλους πυλώνες. Για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θελήσαμε να συμπληρώσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, δουλέψαμε πάνω στον ορισμό της προσθετικότητας. Θεωρήσαμε ότι ο ορισμός ήταν αρκετά γενικός και θελήσαμε να μιλήσουμε για τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης και για το κριτήριο του κινδύνου. Είναι δύο στοιχεία τα οποία θα μας δείξουν κατά πόσο τελικά θα υπάρξει όχι προσθετικότητα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Και θελήσαμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και όσον αφορά τους στόχους, τις πολιτικές και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τη διακυβέρνηση, για το Strategic Board και το Operational Boards. Και δουλέψαμε πολύ και πάνω στο άρθρο 8, το οποίο αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής για τη χρήση της εγγύησης. Μια πολύ γενική ε, μία γινόταν, νομίζω, θέλαμε πιο συγκεκριμένα τους, τέχ, τους στόχους, αλλά και τα scoreboard, το βαθμολόγιο κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θελήσαμε να εφαρμόσουμε όπως έχουμε κάνει και με το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Διευκρινίσαμε περισσότερο και όλο το μήνυμα που έχει να κάνει με την αξιολόγηση και την λογοδοσία και στα πλαίσια της προσθετικότητας. Αλλά επειδή πιστεύουμε ότι θα έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις στα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Θελήσαμε επίσης να ασχοληθούμε και με την ε, δικαιοδοσία των μη συνεταιριστικών ε, δομών. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε λοιπόν την πρόταση με την οποία βασικά συμφωνούμε. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε τους ευρωβουλευτές που σίγουρα με τις παρεμβάσεις τους θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους τρεις συζητητές. Έχουμε τώρα σκιώδεις εισηγητές από τις διάφορες ομάδες. Ξεκινάμε με την κυρία Χάουταλα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Βλέπω ότι υπάρχει σύγκληση μεταξύ των τριών επιτροπών και μεταξύ των τριών εισηγητών. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για αυτή την καλή συνεργασία κατά τους τελευταίους μήνες. Το Ταμείο αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε σε συνδυασμό με τους άλλους δύο πυλώνες του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι μίλησαν για τη σημασία της τεχνικής βοήθειας, που είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να είναι τεχνική βοήθεια. Έχουμε ένα καινοτόμο εργαλείο για την ανάπτυξη, που βρίσκεται σε συνέπεια με τους αναπτυξιακούς μας στόχους. Ιδίως η εγγύηση μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική δύναμη. Έχω τρία ερωτήματα προς την Επιτροπή. Ακούσαμε ότι υπάρχουν εκθέσεις ε, για τα μέσα συνδυασμού των πηγών και δεν ε, είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτά τα συνδυασμένα μέσα. Δεν ξέρω αν έχετε να σχολιάσετε κάτι. Δεύτερον, Δέχεστε την πρόταση των εισηγητών για την εξασφάλιση της προσθετικότητας της χρηματοδότησης και τρίτον μπορείτε να σχολιάσετε σε ποιον θα πρέπει να ανοίξουν αυτά τα κονδύλια σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή και σε άλλους. Ευχαριστούμε. Θα απαντηθούν αργότερα οι ερωτήσεις σας. Στη συνέχεια δίνουμε το λόγο στην κυρία Γιατεμάκη. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη ελέγχθη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα βασικό λόγο για την μετανάστευση. Και δυστυχώς θα συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον ως αιτία μετανάστευσης και γι' αυτό μου είναι δύσκολο να κατανοήσω γιατί δεν έχει τοποθετηθεί η μετανάστευση υψηλότερα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής σε σχέση με αυτό το νέο μέσο. Θα πάρω το παράδειγμα της Συρίας. Η αλλαγή του κλίματος και εκεί βρίσκεται πίσω από τη μετανάστευση. Και βέβαια ο πόλεμος είναι ο πιο σημαντικός παράγων της μετανάστευσης, αλλά και πριν ε, ο πόλεμος εξαναγκάσει τους ανθρώπους να μετακινηθούν. Υφίστατο και ο λόγος της κλιματικής αλλαγής. Άλλο ένα στοιχείο είναι τα χρήματα. Η Επιτροπή προτείνει μόνο 20% των χρημάτων ε, του Ταμείου ΕΤΒΑ να αφορούν την κλιματική αλλαγή. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ως στόχο το 33%. Ο δικός μας στόχος νομίζω θα έπρεπε να είναι το ίδιο, να είναι γύρω στο 35%. Τρίτον, Η πρόταση αυτή θα περικόψει τη χρηματοδότηση της πολιτικής γειτονίας. Μπορεί να είναι λογικό, μεν, αλλά ήδη γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα ούτε καν τώρα. Ερωτώ λοιπόν, θα ήταν δυνατόν να ληφθούν χρήματα από την πολιτική διεύρυνσης γιατί γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό, αλλά επειδή δεν υπάρχουν ε, δράσεις αυτή τη στιγμή σε αυτό τον τομέα λόγω της κατάστασης στην Τουρκία και γενικότερα, μήπως θα μπορούσαμε να πάρουμε χρήματα από την πολιτική διεύρυνση. Αυτές είναι οι τρεις μου παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λόζινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μιλήσω για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το Ταμείο αυτό. Κατά τη σύνταξη της ε, δικής μου έκθεσης για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην αναπτυξιακή βοήθεια ασχολήθηκα και εγώ με, ένα θέμα ότι υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πολλά κράτη-μέλη χρησιμοποιούν ε, πυρογνώμονες και ιδιωτικές εταιρείες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στις χώρες της ανάπτυξης. Η ActionAid υπολογίζει το ποσοστό αυτό στο 81% της αναπτυξιακής βοήθειας ε, που επανέρχεται στις χώρες οι οποίες παρέχουν ενίσχυση. Εδώ μιλάμε για ένα ταμείο εγγυήσεων. Μιλάμε για ε, ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και κατά πόσο είναι βιώσιμος αυτός ο στόχος. Ε, ενισχύουμε την ανάπτυξη στις χώρες στόχο. Τι μηχανισμούς θα μπορούσαμε να βρούμε. Και πώς μπορούμε να βρούμε κάποιους μηχανισμούς ώστε να κατευθύνουμε τα χρήματα αυτά στις ε, ε, αναπτυσσόμενες χώρες, στις χώρες στις οποίες παρέχεται η ανάπτυξη και όχι να ενισχύουμε τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες που είναι οι δωρητές. Επίσης, Σημαντικό είναι ότι υποστηρίζονται προγράμματα καταπολέμησης του αλφαβητισμού, προγράμματα τα οποία θα βοηθούσαν την ε, διαβίωση ε, των πολιτών στις ε, χώρες στόχο και θέλουμε να προάγουμε τη σωστή κοινωνική και οικονομική πολιτική στις χώρες στόχο και επαναλαμβάνω όχι να ενισχύουμε τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες δωρητές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για το επιτελεστέν έργο. Για το κείμενο Σημερίζουμε την υπρασπιστήσα θέση. Θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες, υπενθυμίζοντας κάποια στοιχεία. Το πρώτο, ευρωπαϊκή προτίμηση όσον αφορά την εφαρμογή των μέσων. Δεύτερη τροπολογία, πρέπει να υπάρχει συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Τάπης Επενδύσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση του ταμείου αυτού και θα πρέπει οι αναπτυξιακοί φορεί των κρατών μελών να συμμετέχουν. Τρίτο και τελευταίο σημείο. Εάν χρειαστεί να ανταποκριθούμε στους στόχους της αναπτυξιακής ε, βιώσιμης ανάπτυξης, ε, θα πρέπει να λάβουμε αυτές τις στοιχείες υπόψη. Ευχαριστώ. Ο Σαρλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αυτό το Ταμείο Επενδύσεων είναι έξοχη ιδέα δεν ξέρω γιατί δεν είχαμε πιο πριν αυτή την ιδέα. Διότι αν πάει πολύ καλά, δίνουμε εγγυήσει, αν οι επενδύσει δώσουν αποτελέσματα, δεν αποσύρουμε την εγγύηση. Άρα δεν υπάρχει εκταμείευση, όλα πάνε καλά. Τα ποσά που θα επενδυθούν, αν στοιχηματίσουμε στο μέλλον, οι επενδύσει θα είναι ευφυεί. Αν είναι ευφυεί και συνετέ αυτέ οι επενδύσει, μπορούμε να κάνουμε πολύ, πάρα πολλά πράγματα με ελάχιστα μέσα τα ωφέλη του Ταμείου. Τα πλεονεκτήματα. Επιτρέπει την αντιστροφή των χρηματοπιστωτικών ροών, ενθαρρύνοντας τους επενδυτές, ε, κυρίως τους Ευρωπαίους επενδυτές, τα χρήματα που εγκαταλείπουν τις αναπτυσσόμενες χώρες για να έρθουν σε εμάς τελικά να ακολουθήσουν, να ε, αντισταθμιστούν από τις επενδύσεις που γίνονται στις χώρες. Παράγεται έτσι απασχόληση και έτσι τελικά ταρακουνούμε τους επενδυτές. Λοιπόν, δεν μπορούμε να, κάνει τα πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχουν χρήματα στο ιδιωτικό τομέα. Και στην Αφρική υπάρχουν χρήματα. Οι εταίροι τη Ένωση, τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εμπορικέ τράπεζε, οι επιτόπιε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Αφρικανική Τράπεζα Αναπτύξεω είναι πολύ χρήσιμοι συνεργάτε, διότι η κατάσταση στον αφορά τι πιστώσεις δεν είναι πάντα ίδια στην Αφρική όπω εδώ. Εμεί έχουμε κρίση ρευστότητα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι οι αφρικανικέ χώρε έχουν παρόμοια κρίση ρευστότητα. 12 χώρε απογειώθηκαν, υπάρχουν χρήματα. Έχουν λοιπόν ε, αποταμίευση που πρέπει να κινητοποιηθεί. Για όλου αυτού του λόγου θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα, πάρα πολύ καλή ιδέα. Μετά, δεύτερον, η επιλεξιμότητα βάσει κριτηρίων τη επιτροπή ε, ανάπτυξη του ΩΣΑ. Εκεί δεν έχω κάποια άποψη διότι τα χρήματα που θα επενδυθούν σε αυτό το ταμείο, στο βαθμό που απορροφώνται, δείχνουν αποτυχία. Δεν μπορεί η επένδυση, μάλλον, εάν δεν πάει καλά η επένδυση, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Δεν πετυχαίνουν πάντα επενδύσεις. Η επιλεξιμότητα είναι πιο ευφυής αυτή από την ε, προηγούμενη προσέγγιση. Έχουν δημιουργήσει χρέη πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και μετά η πληρωμή αυτών, πληρωμή αυτών οδηγεί σε εγγραφή στον συλλογισμό των χωρών και γίνονται επιλέξιμες χώρες μέσω αναπτυξιακής βοήθειας. Αλλά περνάνε από τα ταμεία του κράτους τελικά τα χρήματα για να γεμίσουν τις τσέπες κάποιου διαφθαρμένου ηγέτη. Θα πρέπει να σχετικοποιήσουμε τα πράγματα. Αυτή η επιλεξιμότητα δεν θα πρέπει να δημιουργεί πολλά προβλήματα. Λοιπόν, τρίτον, σκέψη αυτή τώρα. οι χώρες που χρειάζονται πιο επίγοντος επενδύσεις είναι αυτές που είναι οι λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές. Εκεί θα πρέπει να παίξει ρόλο εγγύηση. Υπάρχουν περιοχές όπου ακόμα και με τις εγγύησεις δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Αυτό το ολοδιάβημα που δείχνει να είναι περισσότερο τεχνοκρατικής φύσεως. Χρειάζεται πολιτική ηγεσία στεναρή. Και το θέτω το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θα έπρεπε να ετοιμαστεί λίστα συνοδευτικών μέτρων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τι επενδύσεις, να δώσουν καρπούς. Τι εννοώ συνοδευτικά μέτρα. Υπάρχουν χώρες όπου είναι τέτοια διακυβέρνηση όπου κανένας επενδυτής δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο να επενδύσει εκεί θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε τι λόγω χώρε όπου υπάρχει μονίμως κινδύνος και πολύ μεγάλος για να χρησιμοποιηθεί το σύστημα εγγύησεων. Μήπως όπως κάναμε και τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ευρώπη και στο Βέλγιο να έχουμε ειδικέ επενδυτικέ ζώνες ασφαλείς μετά από συνεννοήσεις μεταξύ δικαιούχων χωρών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε να προστατεύονται οι επενδύσεις να κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια. Και αυτή η προσπάθεια μπορεί τελικά να έχει θετική συνέπεια για τη διαχείριση της χώρας. Αυτά ήθελα να πω λίγο πολύ. Ο Ζαν Αρτουί στην αρχή αναφέρθηκε σε έναν ολόκληρο γαλαξία α, κονδυλίων έκτος από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώση που χρηματοδοτούνται και από τα κράτη-μέλη και από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και δημιουργούν πρόβλημα όσον αφορά του ελέγχου. Εξασφαλίζοντα ηγεσία πολιτική που ανταποκρίνεται σε αυτό το τίτλο, μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο διασπάθησης των χρημάτων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει μια κατάλληλη δομή που θα εξασφαλίζει και μια πολιτική κατεύθυνση στον τομέα. Ο κ. Φανσουλίκα εκ νέου, εκ μέρους της Οράγια Post, που είναι σκιώδης της ΑΦΕΤ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνάδελφος επισκέφτεται τη Γενέβη. Έχουμε τρεις αντιπροσωπείες εκεί. Απουσιάζει και μου ζητεί να παρουσιάσει θέση της. Για τους σοσιαλιστές, λέει, το σημαντικότερο θέμα έχει τεθεί στο σχέδιο εκθέσεως, ως έχει. Ως σκιώδη της ΑΦΕΤ, η κυρία Πόστ είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη όσον αφορά τη ρητή αναφορά στο άρθρο 21 των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι σημαντικό να στηρίξει αυτό το Ταμείο την ανάπτυξη και πρόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας, της ειρήνης και του κράτους δικαίου, που είναι ο μόνος τρόπος να αποφευθούν οι συγκρούσεις και να προωθηθεί και να ενισχυθεί η διεθνής ασφάλεια. Όλα αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία όσον αφορά το Ταμείο αυτό, που θα είναι επιτυχές έτσι Αντιμετωπίζοντα τα ριζικά αίτια των μεταναστευτικών πιέσεων. επίση, υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση αυτή καθ' αυτή δεν αποτελεί πρόβλημα. Ο κόσμος θα πρέπει να μπορεί να μετακινείται μεταξύ χωρών αν το επιθυμεί αυτό και αν του αρέσει. Δεν θα πρέπει να υποχρεώνεται να μεταναστεύει λόγω ελλείψης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών για διαβίωση. Συνεπώ, για την κυρία Πόστ και για ε, του σοσιαλιστέ, το ταμείο αυτό το ψηφιακό πρέπει να είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο και εδώ τα ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα των φύλων και κοινωνικό περιβάλλον και ο σεβασμό αυτών των πτυχών είναι στο επίκεντρο. Άλλα σημαντικά θέματα τα οποία έχει θέσει σαν τρίτη κοιόδη που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση είναι η πλήρη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών και των σχετικών οργανώσεων στι διάφορε διαδικασίε που πρέπει να είναι διαφανεί επίση έχει προσθήκε μέσω τροπολογιών. Εν στο άρθρο 21, η μνήμα αυτού του άρθρου είναι καλή, αλλά δεν αρκεί δυστυχώ. Είδαμε από την εμπειρία μα με άλλα ταμεία στο Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την εντολή ότι η αναφορά, η μνήμα του άρθρου 21 δεν σημαίνει αυτομάτω ότι μια αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το πώ επηρεάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται. Θα πρέπει να βάλουμε μια παράγραφο που θα λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα καταρτήσει ένα πλαίσιο και μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση τη συμμορφώσεω με τι επιταγέ του άρθρου 21. Η πτυχή του φίλου αναφέρεται στην έκθεση, αλλά θα ήταν ευνοϊκό αν τονιστεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στην Επιτροπή. Γενική Διευθύνση ΝΙΕΡ. Η κυρία Μαρτίνοβα, παρακαλώ. Δυόμιση λεπτό καθένας, εντάξει. Τρεις ομιλητές έχουμε από την Επιτροπή, δυόμιση λεπτά ο καθένας. Ωραία. Τηλεγραφικά θα τα πούμε κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσουμε. Ματέρνοβα λέγομαι. Πρώτα απ' όλα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ταχύτητα, την επικοδομητική αντιμετώπιση των τριών κοινοβουλευτικών σας επιτροπών. Προσπαθήσαμε και εμείς με τεχνικές συναντήσεις να τη στηρίξουμε. Ανταποκρίθηκαν πάντως πολύ γρήγορα, οπότε ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε που δέχεστε την επέκταση του Ταμείου στο μέλλον και σε άλλες χώρες. Ευχαριστούμε για αυτήν την τροπολογία. Όπως επίσης και τα όσα έχετε διατυπώσει για την προσθετικότητα. Γιατί πιστεύουμε ότι πράγματι είναι κάτι σημαντικό. Από τις συζητήσεις που είχαμε και με τον ιδιωτικό τομέα, δείχνει ότι θα μπορούσε να ήταν κάτι από το οποίο όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Και χαίρομαι για τα σχόλια του κ. Γκέρενς. Ναι, είναι κάτι που θα έπρεπε να είχαμε σκεφτεί νωρίτερα, σύμφωνοι, αλλά πας περιπτώσει τουλάχιστον το έχουμε τώρα. Με την εντολή η ανάπτυξη να πάει από τα δισεκατομμύρια στα 3 εκατομμύρια και για να γίνει αυτό πρέπει να προσελγίσουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Η εγγύηση λοιπόν είναι κάτι από το οποίο ε, μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή και να κερδίσουμε. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέσα που θα επισημάνουμε. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να προετοιμαστεί καλά ε, η δουλειά με διάφορα προγράμματα. Η τεχνική αρρωγή λοιπόν που είναι ο δεύτερος πυλώνας και η τεχνική αρρωγή για τον τρίτο πυλώνα που είναι η βελτίωση επενδυτικού κλίματος είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Μπορεί τεχνικά να μην αποτελούν μέρος της νομοθεσίας που συζητάμε, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο αποτελούν κάτι πολύ θετικό. Τώρα, για τον ιδιωτικό τομέα. Κάνουμε έκκληση για ευελιξία. Πιστεύουμε ότι τα κριτήρια επιλογής που προσθέτουν όλες τις πτυχές που μας ενδιαφέρουν δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχνάμε ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα νέο μέσο με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, Αυτό μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία να έχουμε πάρα πολλά παραρτήματα, πάρα πολλές κατευθυντήριες γραμμές και πολλά σενάρια να ακολουθούμε. Γιατί αυτό μπορεί να τρομάξει κάποιους ε, ιδιωτικούς επενδυτές και να τους απομακρύνει. Το ίδιο ισχύει και με το βαθμολόγιο. Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατικών Επενδύσεων, αυτό μπορεί να λειτουργήσε, γιατί είναι ένα οικονομικό εργαλείο που διαχειρίζεται ένας φορέας. Εδώ όμως έχουμε πολλούς παίκτες και πολύ διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους πυλώνες 2 και 3. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να έχουμε βαθμολόγιο. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την έκκληση. Δείξτε κατανόηση. Δύο πράγματα ακόμα θέλω να πω. Πρώτον, και οι συνάδελφοι φυσικά θα απαντήσουν στα υπόλοιπα για την Ευρωπαϊκή Προτίμηση. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια ανοιχτή πρόταση. Ο λόγος που θέλαμε να παραμείνει ανοιχτό και να συμμετέχουν όλοι είναι γιατί θέλουμε και άλλες πρωτοβουλίες και να γίνει ένας καλός συντονισμός για να είμαστε αποτελεσματικοί. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, για τις συγκρούσεις που τις πλήττουν, τότε δεν υπάρχουν πολλοί παίχτες γύρω τους. Γι' αυτό και θέλουμε να έχουμε την πόρτα ανοιχτή για τη συμμετοχή όλων. Και τέλος για τη διεύρυνση, αν μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα από εδώ, η συζήτηση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και τα θέματα που συζητιούνται για τα Βαλκάνια μάλλον θα μας οδηγούσαν στο να το αρνηθούμε αυτό, να μην το θέλουμε. Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συζητές από τις τρεις επιτροπές αξιότιμα ε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Θέλω, όπω και η Κατερίνα, να σα ευχαριστήσω για τη βελτίωση που βλέπουμε ε, να επιτυχάνετε με ε, τα σχόλιά σα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιε από τις ερωτήσεις. Καταρχήν, όσον αφορά το συνδυασμό των μέσων, μια αξιολόγηση θα δημοσιευθεί κατά τα τέλη Μαρτίου και δεν είναι αρνητική. αντιθέτω. Ε, περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία που μας δείχνουν ότι ήταν ε, σωστό το ότι μετά από 7-8 χρόνια ε, πορείας με την, το συνδυασμό μέσων περνάμε σε μια καινούργια φάση με καλά αποτελέσματα. Η προστατικότητα είναι πολύ σημαντική. Πολλοί από εσά είπατε τι γίνεται όταν ε, δεν γίνονται επενδύσει, όταν είναι πιο δύσκολε οι επενδύσει. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος του επενδυτικού σχεδίου να δώσει μια όθηση και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα καλύτερα κίνητρα και η καλύτερη προπαρασκευαστική εργασία μπορεί να μην επιτρέψει στι επενδύσει να υλοποιηθούν αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και να προσπαθήσουμε και όλα τα συνοδευτικά μέτρα που ανέφερε ο κ. Γκέρενς και άλλοι είναι θεμελιώδους σημασίας και γι' αυτό έχουμε τρεις πυλώνες. Όχι μόνο ο χρηματοδοτικός πυλώνας, αλλά και ένας πυλώνας σχέσεων και διπλωματικός πυλώνας. Και υπάρχει και ο πυλώνας της αναπτυξιακής πολιτικής. Εδώ είναι ο διάλογος με τις κυβερνήσεις, όχι μόνο με την αγορά και τις επιχειρήσεις, αλλά και με τη δικαιοσύνη και με το κράτος δικαίου για θέματα όπως ε, η διαφθορά κλπ. Ο πολιτικός διάλογος λοιπόν, οι πολιτικές πτυχές του διαλόγου είναι εξίσου σημαντικές με τις οικονομικές πτυχές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, αυτές ε, τις τρεις πτυχές, ε, δηλαδή πολιτικές πτυχές, ανάπτυξη πολιτικών και χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό είναι το τέλειο μείγμα το οποίο διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό ε, ε, αναζητούμε λύσεις με ειδικέ επενδυτικές ζώνες κλπ. Δεν υπάρχει μια θαυματουργή λύση για όλα τα προβλήματα, αλλά αυτή η μεταβλητή δημιουργία και ο διάλογος σε κάθε χώρα θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η πολιτική δομή με την οποία διαχειριζόμαστε αυτό το επενδυτικό εργαλείο αποτελεί διασφάλιση του ότι όντως θα τηρηθούν οι στόχοι αυτού του σχεδίου. Θέλουμε η προσθετικότητα των επενδύσεων σε δύσκολες περιοχές, με δύσκολους όρους, να λάβει χώρα και γι' αυτό θα συμμετάσχουν όλοι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όλα τα ευρωπαϊκά μέσα και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν έχουν επαρκείς προτάσεις οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη επενδύσεων, θα καταφύγουμε σε άλλους εταίρους. Αυτή είναι η γενική ιδέα του ότι θέλουμε γύρω από το επενδυτικό σχέδιο να συγκεντρώσουμε ένα αριθμό εταίρων που θα αποδώσουν τα σωστά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φιλιμπέρτο Τσεγιάννο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι συνάδελφοί μου τα είπαν σχεδόν όλα. Uh, να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Καταρχά υποστηρίζουμε ένθερμα πολλέ τροπολογίε και τα σχόλια που ακούστηκαν. Πράγματι, πρέπει αυτό το εργαλείο θα πρέπει να καλύπτει προβλήματα εφράστων χωρών, λιγότερο αντικείμενων χωρών ούτως ώστε να δημιουργηθεί ο κατάλληλος μηχανισμός, κυρίως μέσω δημιουργίας επενδυτικών ευκαιριών για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο κανονισμός δεν μπορεί να είναι πολύ περιοριστικός από αυτού. Στόχος όμως υφίσταται. Πρέπει να επιδιωχθεί και πρέπει να του δοθεί επιχειρησιακό χαρακτήρα στον καθορισμό των ευκαιριών που παρουσιάζονται υπό τη μορφή παραθύρων στο κείμενο για επενδύσει. Ευπρόσδεκτε οι προτάσει περί ενισχύσεω των σημείων περί υπεύθυνη επενδυτική συμπεριφορά, κοινωνική ευθύνη των εταιριών, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμό συμβάσεων και προσανατολισμών που υπάρχουν. Θέλουμε να προωθήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη, που αυτό συνεπιφέρει και πρόοδο στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα. Δεν θα επαναλάβω τα ήδη αναφερθέντα. Είναι πολύ σημαντική η πολιτική διαχείριση του εργαλείου από τις αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και από, τους, τα θεσμικά μας όργανα. Στο τέλος ακούστηκε κάποιο σχόλιο για τον κίνδυνο της διαθέσεως των πόρων που δεν θα πηγαίνουν στις ε, επιλέξιμες χώρες ή θα, και ανταυτού θα επιστρέφουν στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Χρειάζεται και οικονομική διπλωματία όμως τα επενδυτικά σχέδια. Έτσι μπορούμε να παράσχουμε ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη εξαιρετικά προγράμματα στις χώρες αυτές, αλλά και να δημιουργούμε ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και να δημιουργούμε και θέσει εργασία και ευκαιρίε για το τομέα μα, όπω την πράσινη οικονομία, όπου οι ευρωπαϊκέ εταιρείε μπορεί να αγγιθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω, συνάδελφοι, 24 Μαρτίου το μεσημέρι προθεσμία για τι τροπολογίε. Ξανά ο λόγο πάει στον κύριο Αχτουί, ο οποίο λέει, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό μοχλό ανάπτυξη η πρόταση αυτή που εξετάζουμε. Νομίζω ότι θα ήταν ε, καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατυπώσουν συνολικά την πολιτική φιλοδοξία η οποία χρειάζεται ένα τέτοιο εργαλείο. Διότι έχουμε διάφορα μέσα. Σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, για παράδειγμα, αναφερθήκαμε σε αυτό. Ωραία, είναι ενδιαφέρον αυτό που συζητάμε, αλλά δεν το καταλαβαίνει απαραίτητα ο Ευρωπαίος πολίτης, ενώ οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται να καταλαβαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει την προσπάθεια να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να ανταποκριθεί στις ανησυχίες τους, για παράδειγμα, στις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Εξαιρετικά όλα αυτά που περιλαμβάνονται εδώ. Υπάρχει λοιπόν συνεισφορά υπό τη μορφή εγγύσεων, αλλά φοβάμαι ότι δεν φτάνει. Χρειάζεται και προσωπική εμπλοκή επιτόπου στα πλαίσια της συνεργασίας. Και είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ανακοίνωση για ένα συγκεκριμένο εργαλείο χωρίς να διατυπώσει τη συνολική της φιλοδοξία και τα άλλα μέσα που σκοπεύει να διαθέσει στις χώρες που θέλουμε να βοηθήσουμε για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Οπότε, λίγη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς που μας έδωσαν τα 10 λεπτά.